Good afternoon, everybody. We are having a heavy voting session. We are starting with my report on uh, tax. Uh, να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης ε, και της φοροδιαφυγής. Πρέπει να κάνουμε πρώτα βέβαια μια δοκιμή για την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Έχουμε 20 λοιπόν άτομα που ψηφίζουν. Ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση στα αγγλικά πριν να ξεκινήσουμε. Την Παρασκευή στην Όσικτον έλαβε χώρα μια συνεδρίαση της 20 με τους Υπουργούς Οικονομικών και αποφάσισαν ε, ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να είναι κάτι που θα γίνεται συνήθως από εδώ και πέρα και όλα τα κράτη πρέπει να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. Επομένως, ε, έγινε πολύ μεγάλη πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Ήθελα να το δηλώσω αυτό. Έτσι λοιπόν, ε, η δική μας ψηφοφορία δεν θα πρέπει να είναι κάτι πιο οφθοδρομικό σε σχέση με το τι κάνει σήμερα. για ένα συγκεκριμένο τεχνικό θέμα. Έχουμε πάρα πολλέ ψηφοφορίε. Συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπατε, αναρωτιέμαι. Αν, ε, επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ψηφοφορία, αν μπορούμε να δούμε αν έχουμε ομαδικές ε, ψηφοφορίες, να ψηφίσουμε σε μπλοκ κάποια θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, για την τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. 2 και 3 σε μπλοκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 4. Έχουμε ετοιματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ κατά, εποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 5, 6 και 7, υπέρ, κατά εποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 7. 8 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Τμηματική ψηφοφορία. Πετρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10, 11 και 13. Μέχρι και τη 13. Εντάξει, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται από τη 14 18. 15 έως 18 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνονται. 19 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Επιλογή 20 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται και για την γραμματοδότηση του συνολού της όπως υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι, πέρας. Ναι. Ομόφωνη διαθέτηση. Σας ευχαριστώ. Τώρα έχουμε την πολύ σημαντική έκθεση του κυρίου Κασμάρακ. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 και 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογή 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 76, τμήματική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός περιφωνικά υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στο ε, ΦΑΜ 26 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Φάμε 32. Συγγνώμη 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Φάμε 34. Υπέρ. Κατά. αποχες Να αλλάξουμε. για την ΦΑΜ 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισε το όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. και 79. Υπέρ. Κατά. Εποχές. να ελέγξουν. Άρχεται η ψηφορία. το όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 84, υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός 8, τμήματική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εποχές να ελέγξουν Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, εφηγήθηκε και ο συμβασμό 8. Περνάμε στο τροπολείο 89. Υπέρ. Κατά. εποχέ, Εγκρίνεται. Συμβασμό 9. Υπέρ. Κατά. εποχέ, Εγκρίνεται. Για το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Τροπολογία 92 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ...95 και 96 μαζί, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνονται. 97 υπέρ. και 98 εντάξει υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνονται. Συμβεσμός 10 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός υπερφών 11 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη. Το πρώτο τμήμα ψηφίσαμε, περνάμε στο δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο συμβασμό 12. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εντοχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Νομίζω απορρίπτεται. Κατά 8. Λοιπόν, να ψηφίσουμε όλο αυτό για να είμαστε σίγουροι και θα δούμε στη συνέχεια τι θα το τη την γραμματεία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 108. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνει. 110. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται και τον 11 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 112 τμήματική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα Well, I think we the third part of this uh, article. Λοιπόν, να ψηφίσουμε το τρίτο τμήμα. Υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 113. Υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία ΦΑΜ, 3. Υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 φαμ, υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. Τώρα έχουμε τροπολογίες από την Επιτροπή των Γυναικών, 12, υπέρ, κατά, αποχές, συγκρίνεται. 13, υπέρ, κατά, εποχές γκρίνεται. 15 υπέρ κατά εποχές γκρίνεται. 21 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές για να δούμε άρχεται η ψηφοφορία ψήφισα το όλοι πέρας εγκρίνεται Φαμ 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 116-117-118 σε μπλοκ υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 122, 123, 124 μέχρι και την 125 σε μπλοκ, όχι. 122 και 123, υπέρ, κατά. Εποχές εγκρίνονται. 124, υπέρ, κατά. Εποχές εγκρίνεται και τον 25 υπέρ κατά εποχές γκριντ. και τον 26 υπέρ κατά εποχές γκριντ. και τον 27 υπέρ κατά εποχές γκριντ. 128 χωριστή ψηφοφορία πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό 129 και 30 από όχι μόνο 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική λίστα 14 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά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 Λοιπόν, εδώ κάναμε ένα λάθος. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται. Και τώρα πάμε Πάμε στην 137 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 141 υπέρ. Κατά. Αποχές Ας το επαληθεύσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, ας το τσεκάρουμε Λοιπόν, για το δεύτερο τμήμα της 143 άρχεται η ψηφοφορία. Όλοι ψήφισαν εκτός από ένα άτομο. Ωραία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. από την Επιτροπή ΦΑΜ. ΦΑΜ 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 ΦΑΜ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε να το ελέγξουμε Όχι Ωραία Προχωρούμε στο συμβιβασμό 17. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18, συμβιβαστική λύση 18. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 155 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φαμ 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή συμβαστική λίστα 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173 ε, χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ωραία να το ελέγξουμε 173. Πρώτο μέρος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας μάλιστα απορρίπτεται. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. 179 χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική λύση 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, Συγγνώμη, μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο τμήμα, γιατί είναι χωριστή ψηφοφορία που ζήτησαν οι πράσινοι. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. να ελέγξουμε την τελευταία ψηφοφορία. Λοιπόν, συμβαστική λύση 20, δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Ακόμη ένας πρέπει να ψηφίσει. Well, last Τελευταία ευκαιρία πέρα τη ψηφοφορίας. Ωραία, ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Απορρίπτεται με μία ψήφο. 80 και 81 καταπίπτουν 180, 181 πάμε στην 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική λύση 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική λύση 21 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές καλύτερα το υπερληθεύσουμε αυτό το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής λύσης 21 Disclosed. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική ψη, ε, τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται ο προφορική τροπολογία 1 ναι yes. nope. απεσύρθη Il 24 τότε. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν ενενήντα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Yes. So then it is 197. 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 yes. so, compromise 31. Συμβαστική λύση 31 υπέρ α σε δύο σε δύο τμήματα για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Now we have 200 we have uh, yes 203 who is in 203 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική λύση 26, χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Yes. We will, uh, we will vote the following amendments as it was half rejected. Λοιπόν, 211. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 212 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 213 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 217. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται νομίζω. Για να το ελέγξουμε όμως. 217 λοιπόν. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται όντως. «219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». «220-221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Συμβασμός 28 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λοιπόν, για το δεύτερο τμήμα εδώ του συμβασμού 28 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα, όντω. Τελικά. Τρίτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. I don't know 28, δεν θυμάμαι. Εγκρίθηκε. Α, ψηφίσαμε. 2.23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.22 υπέρ. Παρακαλώ. Α, μέχρι και την 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 2.26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 29 Κατά μετά, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα της 29 ε, υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Then we take amendment two... 2.34 υπέρ. Α, χωρίς, συγγνώμη, κατά τη μεταψηφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. ηλεκτρονικό έλεγχο Άρχεται η ψηφοφορία για την 2.35. Πρώτο μέρο, πρώτο τμήμα. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της 235 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη για το δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας, όχι άλλος ένας. Άλλη μια ψήφος. Εγκρίνεται. Την 2.41 μέχρι και την 2.39 ομαδικός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ίσως ομαδικός 2.43 έως 2.47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 2.46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Και την 2.49 μια στιγμή να δω υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται 2.50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.51 υπέρ έχουμε κατά τη μεταψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα της 2.51 υπέρ α καταπίπτει ...2.54 υπέρ. 2.54. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 264 λέει πρόεδρος 264 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από 2,62 έως 2,67 ομαδικός υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται υπέρ αλλά δεν είπε η πρόταση πια κατά αποχές εγκρίνονται. Δύο, εφτά, τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 276 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επιτροπή ΦΑΜ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γυναικών. 14 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για τα εκτιμώντας, για το προήμιο. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, ακαταπίπτει μάλλον. 21 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Χωρίς... Κατά τη μεταμεσχωρητή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Σχόλια εκτός μικροφώνου. 32 έως 34 μαδικός υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνοντα. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική όχι λέει πρόεδρος. Πάμε στην 38. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 λέει πρόεδρος. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Έως 50 ομαδικός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 53 και 54 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 57-59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Παρακαλώ. 59. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας ψηφορίας. Απορριφθείτε. Επιτροπή Γυναικών στο πρίμιο Α. Α, μια μαγική ψηφοφορία. Μάλλον, όχι, ας ψηφίσουμε για την Α υπέρ πρώτα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τη Β τώρα από την Επιτροπή Γυναικών. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στο προημείο σε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προημείο D, δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφορία για παραθέσεις 21 ε, εγκρίνεται. Φαμ 5 υπέρ, επιτροπή δικαιωμάτων των γυναικών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Στο κεφάλαιο 2 στην παράθεση 2, ποιος είναι υπέρ, Σχόλια εκτός μικροφώνου. Ε, από α, 2 ως 6 ομαδικός υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Να πάμε και μέχρι την 9 ομαδικός. 6, 8 και 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Τροπολογία 10. Υπέρ. Με συγχωρείτε. Την 7 δεν ψηφίσαμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 και 13. Μαζί υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνονται και τις 14, 16, 17 και 15 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Οπότε, επί του συνόλου του τροποποιημένου βεβαίω, του συνόλου υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται και ηλεκτρονικός έλεγχος έναρξη ψηφοφορίας. Δύο ακόμη αναμένουν να ψηφίσουν πέρας ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. 20... 20 υπέρ από τις 24. 20 υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαρεκ για αυτό το τόσο σημαντικό έργο για το μέλλον. Θέλετε να πείτε δύο λόγια. Πολύ ωραία. Ναι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάσμαρεκ και να πω ότι μεταξύ της μέρης ημέρας και της ψηφορίας τον Μάιο να σκεφτούμε λίγο με τις πολιτικές ομάδες τι ψηφίσαμε, γιατί ενδεχομένω υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις, κάποια συγκρόμενα, αλληλοσυγκρόμενα κείμενα. Ε, το λεφτό για να στείλουμε ένα συνεκτικό αυτοσυνεπές μήνυμα μέχρι τον Μάιο και ενώψη του Σεπτεμβρίου βεβαίω στην ε, Νέα Υόρκη, της διάσκεψης του Σεπτεμβρίου στην Νέα Υόρκη. Συγχαρητήρια πάντως στον κύριο Κάσμουρεκ η Γραμματεία βεβαίω σε όλου του συμβούλου θα στείλει το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία ε, για να επιβεβαιώσουν ότι όντω ε, σωστά κάναμε ό,τι κάναμε. Σε αυτό, ε, αύριο στιγμή που θα λάβετε βεβαίω, εντό τριών ωρών να το έχουμε πίσω. Κύριε Πρόεδρε, Μίτσελ. ελπίζω να μην παραβιάζω κανένα κανόνα να ζητήσω να μα σερβιστεί και ο καφέ, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα. It would be even better if we served Irish coffee. Και θα ήταν ακόμη καλύτερο αν σερβίραμε και Ιρλανδικό καφέ. Yes, we will on the... Τώρα να ψηφίσουμε επί τη σύσταση σχετικά με την 68η Σύνοδο της Γενική Συνελευσή των Εθνών. Τροπολογία 1. Ναι, όλα σε μπλοκ. Υπέρ. 1 έως 7. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. υπολογείο 8. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 και 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται να ψηφίσουμε επί όλοι τη γνωμοδότηση όπω τροπήθηκε υπέρ, κατά, εποχέ. εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφορία. Λήξη. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια στον συγγετή, τον κύριο Λυσίκ. Τώρα, η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκθεση Γκέρενς, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 2, υπέρ. Σε μπλοκ. Όχι. 2 και 3. Μάλιστα. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εποχέ συγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Εποχέ συγκρίνεται. 4. Από 4 έως την 8, όχι. 4. Υπέρ. Κατά εποχές συγκρίνεται. 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται Τροπολογία 10 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται Δώδεκα. Όχι, δεν είναι δυνατό νομίζω. Δώδεκα. Τμηματική ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Μάλλον καταπίπτει. 12, 13 και 14 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 15 τιμωματική ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές να το ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 15, ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας, πέρας, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 και 17. Πέρ. Κατά εποχές συγκρίνεται. Γκρίνονται. Να ψηφίσουμε το σύνολο της όπω όπως προηγήθηκε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρας 21. υπέρ και δύο αποχές. Our... Συγχαρητήρια για τον εισηγητή. Έχετε το λόγο κύριε Γκέρενς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα φρονήρη χειροκροτήματα και το Μάικλ για ε, αυτή την ε, τόσο σημαντική συνεισφορά που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Να περάσουμε τώρα στην πληροφορία για την ανασυγκρότηση και τον κρατισμό του Μαλή. Do I have that Et après la question. Ah oui. Excuse me, so there is a supplement. Draft question for oral answer. Έχουμε ένα σχέδιο ερώτηση για προφορική απάντηση στην Επιτροπή. Δεν υπάρχουν εδώ τροπολογίε. που είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επίσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Αέρας. Μετά έχουμε και την ίδια ερώτηση για το Συμβούλιο. Δεν υπάρχουν τροπολογίες υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ερώτηση του Συμβούλου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ομόφωνο. Έχουμε το κατάλογο ψηφοφοριών για την ε, ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμό του Μαλή. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Εποχέ συγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. εποχέ, συγκρίνεται. Τροπολογία 30. Τμήματική ψηφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά εποχέ, συγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 και 35. Όχι. 34 υπέρ κατά εποχέ, συγκρίνεται. 35 υπέρ κατά εποχέ, συγκρίνεται. 36 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται Προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Μάλιστα. Τροπολογία 40 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται 41 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 2 Μάλλον τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 ηλεκτρονικό έλεγχο Άρχεται η ψηφοφορία. Άλλο μία ψήφο. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Την ψηφορία. Καταπίπτει. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, χέρι εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, χέρι εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, χέρι συγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, χέρι συγκρίνεται και τροπολογία τέσσερα. Περνάμε στην τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται 55 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται 56 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται προφορική τροπολογία 5 τροπολογία 57 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 60 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Λοιπόν, να ψηφίσουμε τα εκτιμώντα, τροπολογία 1. Μπορούμε να δούμε σε μπλοκ το 1, 2, 3. Υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Συμβιβασμό 6. Υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 7, υπέρ. Κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 7 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβασμό 4 υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε για το συμβιβασμό 4 άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβασμός 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 και 16 όχι 15 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 5 υπέρ κατά απόχέ <coughs> εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 21, τμήματική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να δούμε σε μπλοκ από την 24 έως και την 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ του ψηφίσματος αυτού. Έτσι όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Unanimously. And, uh, yes, and felicitation from... Συγχαρητήρια για τον εισηγητή. Λοιπόν, προχωρούμε στην έκθεση της Μισελ Στρίφλερ για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών. Η τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 Κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. 15 και 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ομπλουά 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και πάλι από την Επιτροπή Απασχόλησης 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Ομπλουά 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Και άλλη μια ψήφο χρειαζόμαστε, ωραία. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Amendment 1. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. Αμπλουά 14 υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Απασχόληση 15 υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται. Απασχόληση 16 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ε απορρίπτεται τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόληση 17 κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα καταπίπτει θα ψηφίσουμε λοιπόν για το δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επιτροπή Προπολογισμού καταπίπτει. Προφορική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 18. Καταπίπτει. Προπολογισμό, 9. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Απασχόληση 19. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Μάλλον 20 και 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. «22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 καταπίπτει Απασχόλης 21. Απασχόληση 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμός 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 25 και αμπλουά 23 και budget 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και οι τρεις. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Προφορική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 60. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πασχόληση 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30-31 και 30-31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται απασχόληση 28 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμός 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32, 33, 34, 35, yes. υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Απασχόλης 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμός 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόλης 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 37 34. Ε, απασχόληση 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόληση 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απασχόληση 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Απασχόληση 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 και 39 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Απασχόληση 38 κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 39 υπέρ κατά αποχές. να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, 39. Ε, αυτό ελέγχουμε. Και άλλη μια ψήφος. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες τότε. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόληση 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος Κάποιο Κάποιος έφυγε από την αίθουσα αλλά άφησε την κάρτα του εδώ. Λοιπόν, πέρα τη ψηφοφορία απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απασχόλη 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απασχόλη 42. Κατά τμήματα ψηφοφορίας τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ anymore. so, so in favor, uh, yes, so this, donc, I, I want to say maybe in French. Uh, qui, yes. So who is in favor of the third part? Ποιος είναι υπέρ του τρίτου τμήματος, ποιος είναι κατά, αποχή, Απορρίπτεται και το τρίτο τμήμα. Άρθρο 17 πάμε τώρα. Okay. So 42 till 45. 42-45 τροπολογίες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Προπολογισμός 17. Α, και τροπολογία 48 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Προπολογισμός 18. I don't understand. Can we work the second part? Only the second part. Okay. Well, I trust the Secretariat. They say Έχω εμπιστοσύνη στην ε, γραμματεία. Λοιπόν μου λέει για τον προπολογισμό 18 ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 λέει πρόεδρος «47 και 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται». Τροπολογία 51. Η 50 καταπίπτει. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 ως 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Αιτιολογικές σκέψεις. 56 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Προφορική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα πέντε τέσσερα και τρεις μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Προφορική τροπολογία 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απασχόληση 6. Μέχρι την προφορική 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Απασχόληση 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 έως 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9. 10, 11, 9, 9 μόνη της. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία, να ελέγξουμε την 9. Ψηφίστε για την 9. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. δέκα, δέκα έντεκα μάλλον, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Προπολογισμός επτά, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε για την απασχόληση 10. ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Γλωσσική διόρθωση. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα για την έκθεση στο σύνολό τη Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ας το κάνουμε και ηλεκτρονικά για το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με ισοπαλία. 21-21. Έχουμε και δύο ακόμη τροπολογίες από την Επιτροπή Προπολογισμού. Ένα-δύο, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συνεχίζουμε. Προπολογισμό 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου στο σύνολό του. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. με βάση τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν μπορούν να ξεκινήσουν άτυπες διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι, διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι υπέρ. Α, πρέπει να γίνει η ηλεκτρονική ψηφοφορία εδώ. Λοιπόν, ωραία. Με βάση αυτές τις τροπολογίες λοιπόν λέμε να ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας είκοσι ψήφοι περ μία αποχή ουδής κατά οπότε εγκρίνεται και όσον αφορά τη διαπραγματευτική ομάδα πρόεδρος εισηγητής και ένας σκιώδης εισηγητής από κάθε πολιτική ομάδα. Λοιπόν, ψηφίζουμε από αυτού ηλεκτρονικά. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. μία ψήφοι υπέρ, ουδής κατά ομόφωνα υπερψηφίζεται τελειώσαμε με τις ε, ψηφοφορίες χαρητήρια στη Μισελ Στρίφλερ για την έκθεσή της yes. well, δεν έχουμε κάτι στα διάφορα επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 27 Μαΐου και Τρίτη 28 Μαΐου. Σας υπενθυμίζω ότι θα αποδεθούμε και τον Επιτροπό μας. Παρακαλώ να είστε εδώ, γιατί επαναλαμβάνω θα είναι εδώ ο Επίτροπος 28 Μαΐου το απόγευμα. Να είστε όλοι εδώ. Και τώρα θα συνδυάσουμε από κοινού με την ΑΦΕΤ για ανταλλαγή απόψεων με τον Επιτροπό για την κατάσταση στην Συρία και τις επιπτώσεις ε, λόγω των προσφύγων σε Ιορδανία και Λίβανο. PHS 3 σε 50. Εκεί θα συνηθούμε. Στο πενηθήριο 3 σε 50. de place.